ολοκληρώσαμε αυτό το σημείο και πάμε στη δήλωση της Επιτροπής για την πολιτική κατάσταση στην Ονδούρα εν ώψη των εκλογών στη χώρα. Το λόγο έχει. Ας αφήσουμε τους επιτρόπους να φιληθούν. Το λόγο λοιπόν έχει η Επίτροπος Άστον. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, θα συζητήσουμε σήμερα την... τις εξελίξεις της Στην Ονδούρα, με συγχωρείτε. Ναι, τέσσερις μήνες μετά τις εκλογές του Πρόεδρου της δυστυχώς η κρίση εξακολουθεί να μην έχει επιληθεί παρά την συμφωνία της 30ης Οκτωβρίου από την Επιτροπή που εκπροσωπεί τον Πρόεδρο και την de facto κυβέρνηση. Η εφαρμογή της λεγόμενης συμφωνίας του Σαν Χωσέ θα πρέπει να δημιουργήσει ένα πλαίσιο αποκατάστασης της δημοκρατίας και της συνταγματική τάξης στην Ονδούρα, αλλά δυστυχώ δεν είχαμε πρόοδο από την κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας και η κυβέρνηση αυτή απορρίφθηκε από τον πρόεδρο Ζαλία. Επιπλέον το Κογκρέσο ακόμα δεν αποφάσισε ε, να τον αποκαταστήσει στην κυβέρνηση οπότε αμφισβητούνται οι εκλογές 29 ε, της Νοεμβρίου που θα αποτελέσουν το βασικό στοιχείο έξοδου από την κρίση. Οπότε εμείς ζητήσαμε από όλα τα μέρη να εφαρμόσουν άμεσα όλα τα στοιχεία της συμφωνίας ως προϋπόθεση για να επανέλθουν οι σχέσεις μας στα φυσιολογικά πλαίσια συμπεριλαμβανομένης αναπτυξιακή βοήθειας. Η Κομισιόν σήμερα υποστήριξε, μέχρι σήμερα υποστήριξε πλήρως τι προσπάθειες ε, διαιτησία του Πρόεδρου της Κωνσταντίνα, του Σκαλερίας και του Οργανισμού Αμερικανικών Κρατών και τα μέτρα που έλαβε η Διεθνή κοινότητα για να ασκηθεί πίεση στα μέρη για να βρεθεί μια ειρηνική λύση. Ο επιτόπου της Προεδρίας της Ένωσης ανακλήθηκε για διαβουλεύσεις και όλοι οι υπόλοιποι πρέσβεις ε, αποχώρησαν από τη χώρα, η πρέσβεις της Ένωσης. Έχει σταματήσει η συνεργασία ε, όσον αφορά την κοινωνική χρηματοδότηση πλην, τη χρηματοδότηση, πλην της χρηματοδότησης της κοινωνίας των πολιτών Επλέον, Η αποστολή παρατήρηση των εκλογών της 29ης Νοεμβρίου ακυρώθηκε. Παίρνουμε λοιπόν πολύ σοβαρά αυτή την κρίση καθώς είναι ένα βήμα προς τα πίσω για τη δημοκρατία, όχι μόνο για την Ονδούρα και την υπόλοιπη Κεντρική Αμερική, αλλά για ολόκληρη τη Λατινική Αμερική. Θέλω να επαναλάβω πως η Κομισιόν θα υποστηρίξει την ομαλοποίηση της πολιτικής κατάστασης στην Ονδούρα και γι' αυτό χρειάζεται να τηρήσουν τα μέρη την συμφωνία αν και λόγω του περιορισμένου χρόνου δεν είναι πλέον δυνατόν να αποσταλεί αποστολή παρατήρησης εκλογών, στείλαμε δύο εμπειρογνώμονες που αποσπάστηκαν στην ε, τοπική αντιπροσωπεία της Κομισιόν με εντολή να βοηθήσουν στη διεξαγωγή των εκλογών και να συμβουλεύσουν για πιθανή δράση μετά τις εκλογές. Εάν το επιτρέψει η πολιτική κατάσταση θα υπάρξει πιο ενεργή εμπλοκή και η Κομισιόν έχει προβλέψει οικονομική στήριξη για το εκλογοδικείο με μια σύμβαση με το αναπτυξιακό πρόγραμμα του ΟΗΕ. Επίσης είμαστε έτοιμοι να δώσουμε οικονομική στήριξη στον Οργανισμό Αμερικανικών Κρατών εάν προκύψει, προκύψουν προϋποθέσεις για παρατηρητές των εκλογών. Συνεχίζουμε λοιπόν να υποστηρίζουμε κάθε προσπάθεια για να επανέλθει η δημοκρατία στην Ονδούρα. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Περνάμε στις πολιτικές ομάδες για το ΕΛΚ για δύο λεπτά. Ο κύριος Πέτερλε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, αδίτη συνάδελφοι. Πριν από ένα μήνα είχα την ευκαιρία να διαπιστώσω αυτοπροσώπως την κατάσταση στην Ονδούρα. Ήμουν μέλος της αντιπροσωπείας του ΕΛΚ. Επισκεφτήκαμε τον πρόεδρο της Ρίκας, τον κύριο Αρίας και μας παρουσίασε την συμφωνία του Σαν Χωσέ. Συναντηθήκαμε και με τον πρόεδρο Μισελέτη, με τον Υπουργό Εξωτερικών, με δικαστές ε, του συνταγματικού δικαστηρίου καθώς και με υποψήφιους ε, προέδρους και με λοιπούς σημαντικούς εκπροσώπους ε, χαιρέτησαν την αποστολή μας και είναι και οι δύο πλευρές έτοιμες για διάλογο. Νομίζω πως είναι σημαντικό να διασφαλίσουμε ε, το οποίο λέει ο πρόεδρος Ζελά για να μην υπάρξει βία. Και συμφωνούμε με αυτό το οποίο πρότεινε ο πρόεδρος Αρίας. Πρέπει να επιμείνουμε να καταλήξουμε σε μια πολιτική συμφωνία οι εκλογές 29 Νοεμβρίου δεν είναι αποτέλεσμα πολιτικών αλλαγών είχαν ήδη προβλεφθεί αυτές οι εκλογές επί Προέδρου Ζελάγια. Μετά τα γεγονότα του Ιουνίου δεν είχαμε άλλους ε, προ... υποψήφιους Προέδρους γιατί λένε πως ε, δεν θέλουν να επιτείνουν την κρίση και βέβαια είναι πάρα πολύ σημα... μεγάλη σημασία των εκλογών. Η Ονδούρα είναι μια χώρα της Νοτιού Αμερικής με την οποία θέλει να συνάψει μια συμφωνία η Ευρωπαϊκή Ένωση και τώρα σταμάτησαν οι διαπραγματεύσεις. Οι πολιτικές αυτές εξελίξεις ενδιαφέρουν πάρα πολύ την Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό εγώ προτείνω να αποστείλουμε αποστολή παρατήρηση. Σας ευχαριστώ για δύο λεπτά. Κύριος Γιάννης για τους Σοσιαλιστές και Δημοκράτες. Ναι. Πρόεδρε, αφού άκουσα την Επίτροπο, Θα ήθελα να πω ότι σπάει ένας κύκλος μη πραξικοπημάτων 12 ετών στην Λατινική Αμερική με το πραξικόπημα στις Ονδούρες. Δεν μπορούμε να μείνουμε άφωνοι και αδρανείς. Θα πρέπει να υποστηρίξουμε τη διαμεσολάβηση Αρίας και βεβαίως να αξιοποιήσουμε την ομπρέλα του ΟΗΕ. Και να μπορέσουμε να αποκαταστήσουμε τη δημοκρατία. Η νέα κυβέρνηση δεν έχει καμία αξιοπιστία και τα αποτελέσματα των εκλογών δεν μπορούν να αναγνωριστούν από τη διεθνή κοινότητα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αν αποστείλει αποστολή παρατήρηση των εκλογών θα διαπράξει μεγάλο σφάλμα. Θα είναι σαν να αναγνωρίζουμε το αποτέλεσμα του προξικοπήματος. Είμαστε εγγυητής της ελευθερίας, της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Όπω είπε ο Βάκλαβ Χάβελ, δεν μπορούν να υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά. Είμαστε όλοι δημοκράτε. Και ω εκ τούτου υπέρ τη ελευθερία. Είτε Κούβα, είτε Κίνα, είτε Ονδούρα, η στάση μα θα πρέπει να είναι η ίδια. Υπέρ τη ελευθερία, υπέρ τη δημοκρατία, χωρί ιδεολογικού χρωματισμού. Δεν υπάρχουν καλοί και κακοί πραξικοπηματίε. Δεν υπάρχουν αριστεροί και δεξιοί πραξικοπηματίες. Όλοι οι πραξικοπηματίες είναι πραξικοπηματίες και ως τέτοιους θα πρέπει να τους αντιμετωπίσουμε. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ. Για ένα λεπτό η κυρία Μπιλμπάο. Ευχαριστώ πολύ πρόεδρε. Στις 30 Οκτωβρίου υπογράφει η Συμφωνία του Σαν Χωσέ και τα μέρη αποφάσισαν να δημιουργηθεί μια κυβέρνηση εθνικής ενότητας το Νοέμβριο και να επιστραφεί η εξουσία στον πρόεδρο Ζελάγια. Όμως ο κύριος Μιτσελέτε προσπάθησε να δημιουργήσει η κυβέρνηση ενότητας χωρίς τη συμμετοχή του κύριου Ζελάγια. Το Κογκρέσο ψήφισε να μην ε, του επιτραπεί η πρόσβαση στην εξουσία. Ο δεν συμμορφώθηκε με τη συμφωνία, προκήρυξε εκλογές και οι υποψήφοι αποσύρονται διότι θεωρούν ότι δεν πληρούνται οι δημοκρατικές προϋποθέσεις για να λάβουν χώρα οι εκλογές. Επίσης, βία λαμβάνει η χώρα. Σήμερα δολοφονήθηκε ένας ε, ε, δήμαρχος της αντιπολίτευσης και ο σωματοφυλακάς του. Υποστηρίζουμε τις ε, εκδηλώσεις που γίνονται. Υποστηρίζουμε την πρωτοβουλία Λούλα και τη διαμεσολάβηση των ΙΠΑ, αλλά βεβαίως και του διαμεσολαβητού Αρίας. Ζητούμε συμμόρφωση με τη συμφωνία, επιστροφή του κυρίου Ζελάγια στην εξουσία και την αρμονική συμβίωση των κατοίκων της χώρας. Ανάκαμψη του διαλόγου Κάτι το οποίο βεβαίω όλοι συμφωνούμε ότι γίνεται κάθε φορά και πιο δύσκολο. Θα πρέπει και η Ευρώπη να ασκήσει πίεση στους πραξικοπηματίες, ούτω ώστε να διευκολυνθεί η εξέβρεση συμφωνίας. Ζητώ συγγνώμη που περεύει το χρονικό όριο και σας ευχαριστώ για τη γενοδορία σας. Το λόγο έχει τώρα εξ των Πρασίνων για ένα λεπτό η κυρία Γκρέσε. Κυρίες και κύριοι βουλευτέ, μετά από στρατιωτικό πραξικόπημα και την καθαίρεση του νομίμου Προέδρου, η συμφωνία του Σαν Χωσέ θα μπορούσε ίσως να θεωρηθεί σαν καλή είδηση, αλλά δεν υπάρχει πια τέτοια ελπίδα. Οργάνωσε ο ίδιος μια κυβέρνηση εθνικής ενότητας και ο πραξικοπηματίας Μικελέτη συνέχισε να ασκεί την παράνομη δραστηριότητά του και τον αυταρχισμό του. Πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να καταδικάσει όλα αυτά και αμέσως να ζητήσει την παρέτησή του και την επιστροφή του νόμιμου Προέδρου. Δεν μπορούν να οργανωθούν εκλογές από παράνομη δικτατορία. Οι εκλογές της 29 η Νοεμβρίου δεν θα αναγνωριστούν. Όπως και η οργάνωση των Αμερικανικών κρατών και εμείς πρέπει να αρνηθούμε να στείλουμε παρατηρητές και δεν θα λάβουμε υπόψη τα αποτελέσματα τέτοιων ψευτοεκλογών. Είμαστε πολύ ανήσυχοι μπροστά σε τόσες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που μαθαίνουμε. Πρέπει η Ευρώπη να επιμείνει στη δημοκρατία και να αρνηθεί κάθε συμφωνία με μια παράνομη κυβέρνηση. Αν συνεχιστεί δε η σύραξη πρέπει να υπάρξει και παρέμβαση. Έχουμε την ευθύνη να διασφαλίσουμε εκατομμύρια κάτοικοι της Ονδούρας να μπορέσουν να διαβιώσουν δημοκρατικά και να μην δεχτούν το προνομτσιαμιέντο. Ευχαριστούμε κυρία Γκρέσ. Παρόλο που και εσείς ε, που δεν ζητήσατε συγγνώμη προς η κυρία Μπιλμπάου, είστε συγχωρεμένοι. Για ένα λεπτό ο κύριος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 okay. Υπάρχει πρόβλημα με τη διερμηνία, αλλά σε λίγο θα διορθωθεί. Be so kind to start okay. again, please. Eh, eh, Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, εκτιμώ βεβαίω τον συνάδελφο, έχω παρακολουθήσει τα διοδρομία του, αλλά δεν μπορώ να συμφωνήσω με αυτά τα οποία είπε όταν ανέφερε τα λόγια του Προέδρου Χάβελ. Εγώ ήμουν ένας από τα εκατομμύρια που βγήκαν στους δρόμους όταν έβγαζε λόγους ο κύριος Χάβελ. Ήμασταν στον δρόμο, εγώ ήμουν 18 χρονών τότε και θέλαμε ένα πράγμα μόνο. Ε, να, ανεξαρτήτως πολιτικής τοποθέτησης. Θέλαμε ελεύθερες εκλογές. Αυτό νομίζω ήταν ε, το σημαντικότερο και αυτό μας ένωνε όλους όταν λέμε τις εκλογές αυτό σημαίνει δημοκρατία η κατάσταση στην Ονδούρα λοιπόν δεν είναι απλή και ε, εμεί από ε, την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορούμε να το λύσουμε πρέπει να το δούμε αυτό σε ένα ευρύτερο πλαίσιο και νομίζω πως οι εκλογές είναι ένα καλό πρώτο βήμα και πρέπει να στείλουμε μια αποστολή παρατήρηση των εκλογών. Για την ε, Ενωμένη Πράσινη Αριστερά και Βόρεια Πράσινη Αριστερά. Η κυρία Φιγκορέδο. Ευχαριστώ. Στις 28 Ιουνίου στην Ονδούρα το πραξικόπημα αποτέλεσε την τελευταία στεγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι της καταστρατήγησης της συμφωνίας. Είναι απαράδεκτο οι πραξικοπηματίες συστηματικά να αναβάλουν την επιστροφή του Προέδρου Ζελάγια που συνταγματικά είναι ο εκλεγμένος Πρόεδρος της χώρας. Αυτό είναι απαραίτητη και ανεφόρον προϋπόθεση. Χωρίς την επιστροφή του Πρόεδρου Ζελάγια δεν μπορεί να λάβουν χώρα εκλογές. Δεν πληρούνται οι ελάχιστες προϋποθέσεις που θα δώσουν τη δυνατότητα στους πολίτες να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα χωρίς πιέσεις, ανώνυμα, ελεύθερα και κατά συνείδηση. Γι' αυτό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να καταδικάσει απερίφραστα την τακτική των πραξικοπηματιών. Να απαιτήσουμε άμεση επιστροφή της δημοκρατίας και να μην αποστείλουμε παρατηρητές για τις ψευτοεκλογές αυτές. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Φιγκερίδο. Για δύο λεπτά ο κύριος Κασμάρεκ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε κυρίες και κύριοι. Οι εκλογές μπορεί να αποτελούν διέξοδο από το αδιέξοδο. Αυτή ήταν η κατάσταση στην Ευρώπη στο παρελθόν, να θυμηθούμε το 1989 στην Πολωνία. Αλλά οι, εκλογή, οι εκλογές αυτές δεν ήταν δημοκρατικές, ήταν αποτέλεσμα πολιτικού συμβασμού. Δεν ήταν δημοκρατικές εκλογές, ε, ήταν κάτι το ιδιαίτερο όμως και πολύ σημαντικό, αλλά για να είναι τόσο σημαντικές και ιδιαίτερε εκλογέ πρέπει να ε, πληρούν ορισμένου όρου, δηλαδή να τηρηθούν οι πολιτικές συμφωνίες ε, για την οργάνωση αυτών των εκλογών. Κανονικά προκύπτει το πρόβλημα ερμηνείας ε, των συμφωνιών και μετά προκύπτουν διαφορές στην ερμηνεία. Για να μην οδηγηθούμε λοιπόν σε σύγκριση ε, πρέπει να υπάρχει κάτι πολύ απλό αλλά και δύσκολο ταυτόχρονα. Καλή θέληση από τις δύο πλευρές της ε, σύγκρουσης στην Ονδούρα εδώ πέρα συγκεκριμένα. Χωρίς λοιπόν καλή θέληση και από τις δύο πλευρές δεν θα γίνουν οι εκλογές ή δεν θα εκπληρώνουν τις ελπίδες ε, των ανθρώπων. Γι' αυτό εγώ ζητώ καλή θέληση υπευθυνότητα καθώς στο παρελθόν η Ζελάγια και η Μιτσελέτη έχουν κάνει πολιτικά σφάλματα. Οι εκλογές αποτελούν ευκαιρία να διορθώσουμε τα λάθη του παρελθόντος. Και αυτό νομίζω είναι κάτι το οποίο πρέπει να επιθυμούμε γιατί μπορούν να είναι θετικές οι εκλογές. Η Ευρωπαϊκή Ένωση υποστηρίζει αυτή τη διαδικασία και είμαστε ικανοποιημένοι με αυτό. Γιατί, γιατί πιστεύουμε πως η δημοκρατία είναι μία αξία θετική. Ακούστηκε σήμερα σε αυτή την αίθουσα πως ε, πρέπει να κοιτάξουμε το κακό στα μάτια, γιατί αυτό θα εκμεταλλευτεί κάθε αδυναμία μας και η κατάσταση αυτή στην Ονδούρα είναι προσωρινή. Και δεν μπορεί να διαρκέσει για πάντα. Θεωρώ λοιπόν πως οι εκλογές αυτές είναι μια ευκαιρία για αλλαγή. Σας ευχαριστώ για δύο λεπτά η κυρία Μποσκούρτ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε τη 28 Ιουνίου ανετράπη ο πρόεδρος Ζελάγια από, το, από τον στρατό. Το στρατιωτικό αυτό πραξικόπημα καταδικάστηκε εντονότατα. Πρέπει να αποκατασταθεί η δημοκρατική τάξη στην Ονδούρα και με ειρηνικό τρόπο να οδηγηθούμε σε διάλογο. Εδώ και μήνες γίνονται έντονες διαπραγματεύσεις και τυχαία πριν από ε, δύο εβδομάδες όταν τυχαία ήμασταν με την αντιπροσωπεία στην Κεντρική Αμερική είχαμε μια ιστορική συμφωνία που θα σημάνει την αποκατάσταση της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου την αποκατάσταση του εκλεγέντος Προέδρου και της Εθνικής Ενότητας. Μία συμφωνία η οποία αν εφαρμοστεί θα δημιουργήσει νομιμότητα και για τις εκλογές. Η συμφωνία αυτή αυτή τη στιγμή δεν εφαρμόζεται, οπότε θα πρέπει να επιστρέψουν οι δύο πλευρές στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για να πραγματοποιήσουν αυτή την συμφωνία για να αντιστραφεί το στρατιωτικό πραξικόπημα. Αυτή είναι η υποχρέωσή τους έναντι του πληθυσμού της χώρας του. Στην περίπτωση στην οποία δεν έχουμε δημοκρατική λύση, φαίνεται πως αυτή τη στιγμή δεν θα αναγνωριστούν οι εκλογές. Αυτό θα έχει ευρύτατες συνέπειες για την Νότιο Αμερικανική ε, διαδικασία ολοκλήρωσης, καθώς θα έχουμε καθυστερήσεις ετών στην Συμφωνία Σύνδεσης. Τώρα για τους ε, συναδέλφους μου που λένε πως πρέπει να αναγνωρίσουμε τα αποτελέσματα των εκλογών. Έχω να πω το εξής, δεν πρέπει να στείλουμε μήνυμα στην Ονδούρα, την Κεντρική Αμερική και τον υπόλοιπο κόσμο πως εγκρίνουμε την ε, βία. Πρέπει να στείλουμε αυτή τη στιγμή το μήνυμα και αν δεν το κάνουμε αυτό ούτε ο Ζελάγια ούτε ο Μικελέτη θα κάτσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και θα παίξουμε έτσι το παιχνίδι των αντιδημοκρατικών δυνάμεων. Σας ευχαριστώ, ευχαριστώ κυρία Μποσκούρτ. Τον λόγο για ένα λεπτό έχει ο Βίλι Μάιερ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κυρία Επίτροπε, θα ήθελα να σας συγχαρώ και εσάς και την Κομισιόν και το Συμβουλίο διότι επιτύχατε ομοφωνία στα πλαίσια της διεθνής κοινότητας για απερίφραστη καταδίκη του προεξικοπήματος στην Ονδουρά οποιαδήποτε διεθνής ε, παρέμβαση θα ε, ε, περνάει από απαραίτητη προϋπόθεση την επιστροφή του Πρόεδρου Σελάγια. Λυπούμε, λυπούμε βαθέως που το Κοινοβούλιο αυτό δεν έχει ακόμα καταδικάσει το πραξικόπημα. Και δακτυλοδεικνύω τον υπεύθυνο που δεν είναι άλλος από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Είναι απαράδεκτο το κοινοβούλιο αυτό να μην έχει κατοδικάσει το στρατιωτικό πραξικόπημα. Συμφωνώ ότι δεν θέλουμε παρατηρητές, να αποστείλουμε παρατηρητές. Δεν θέλουμε να αναγνωρίσουμε τα αποτελέσματα του Νοεμβρίου, διότι δεν είναι δημοκρατικές α, εκλογές. Με πρόεδρο δημοκρατικά εκλεγμένο, εχμάλωτο στη βραζιλιανή πρεσβεία. Ο κύριος Ιτουργάιτ. Για ένα λεπτό. Ευχαριστώ θα ήθελα ορισμένες ομιλίες για αυστηρότητα κατά της Ονδούρας που έχουν ορισμένοι αριστερών συνάδελφοι να το κάνουν και για τα όσα γίνονται στην Κούβα και για τα όσα κάνει ο Τσάβες στη Βενεζουέλα διότι το τείχος του Βερολίνου, τα γκούλαγκ του Στάλιν ε, είναι καλά και τους βοηθούν παρά οι δημοκρατικές εκλογές όπως στην Ονδούρα τώρα. Και τούτου λεχθέντος θα πρέπει να σκεφτούμε το εξής. Τι έγινε σε αυτήν την κεντροαμερικανική χώρα. Στην Ονδούρα οι προεδρικές εκλογές είχαν ε, προκηρυχθεί εδώ και 16 μήνες. Οι εφορευτική επιτροπή ούτως υπήν. Οι εισαγγελείς που διορίστηκαν για την διεξαγωγή των εκλογών ε, διορίστηκαν ε, ήδη επί Ζελάγια πριν από 16 μήνες. Έγινα ε, πρώτος γύρος. Οι περισσότεροι υποψήφοι θέλουν να γίνουν οι εκλογές στην Ονδωρά. Άρα σε τι βασίζονται ορισμένοι για να μην αναγνωρίσουν την εκλογική διαδικασία. Είτε είναι ο Ζελάγια είτε δεν είναι στην εξουσία. Στις 30 Οκτωβρίου οι διαπραγματευτές και των δύο ε, μερών δεσμεύτηκαν να εξεύρουν λύση για διέξοδο από την κρίση. Υπήρχαν μέτρα που υποστηρίζαν και οι δύο πλευρές οι εκπρόσωποι του έκπτωτου του Προέδρου Σελάγια δεν ήθελαν να προσυπογράψουν τη Συμφωνία για Κυβέρνηση εθνική ενότητα. Οπότε <laughs> είναι σαφέ ότι οι λοιπές δημοκρατικέ δημοκρατικές δυνάμεις θέλουν να προκηρυχθούν και να γίνουν εκλογές με παρατηρητές που θα στείλουμε και η ομάδα μας θα έχει όπως ζήτησε ο διαμεσολαβητής πρόεδρος της Κώστα Ρίκα, Όσκαρ Άρια. Το ίδιο το ίδρυμα Όσκαρ Άρια είχε πει ότι θα αποστέλει παρατηρητές στην Ονδούρα. Θα το κάνουμε λοιπόν, θα στείλουμε παρατηρητές επειδή μόνο και μόνο το ζητάει ο Όσκαρ Άριας. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ. Για ένα λεπτό. Ο κύριος Σόνικ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Νομίζω ότι οι εκλογές της 29ης Νοεμβρίου θα είναι μια ευκαιρία για την Ονδούρα και είναι καθήκον μας να στείλουμε παρατηρητές στις εκλογές αυτές. Όχι με σκοπό να τους, να τους προσδώσουμε νομιμότητα, αλλά για να δούμε πώς θα διενεργηθούν. Εξάλλου Πολύ κοντά εκεί βρίσκεται και η Κούβα όπου δεν έγιναν εκλογές για 50 χρόνια και οι κομμουνιστές εκεί πέρα φυλακίζουν τον κόσμο χωρίς δίκη. Πολλές φορές έχει ζητηθεί απελευθέρωση των πολιτικών εχμαλώτων. Δώσαμε και βραβείο Σαχάροφ σε κάποιον από αυτούς και δεν μπόρεσε, δεν είχε τη δυνατότητα να έρθει να το παραλάβει. Θα ήθελα λοιπόν η αριστερά καθώς και το Συμβούλιο και η Επιτροπή να σκεφτούν και τη, τα δημοκρατικά δικαιώματα των κουβανών. Ευχαριστούμε κύριε Σόνικ. Και τώρα για ένα λεπτό ο κύριος Κόρτες. Πρόεδρε, συνάδελφοι, θέλω να εκφράσω την άκρα ανησυχία μου για την αναστολή της συμφωνίας του Σαν Χωσέ η Ευρω-Λατινοαμερικανική πολέμου χώρα των Παναμά στα τέλη Οκτωβρίου επανέλαβε ότι καταδικάζει το στρατικό πραξικόπημα και υποστηρίζει τις προσπάθειες διαμεσολάβησης. Θα πρέπει να ανανεώσουμε την έκκλησή μας για διάλογο. Η κατάσταση είναι κρίσιμη στην Ονδωρά, όχι μόνο πολιτικά, αλλά κοινωνικά και οικονομικά. Φτώχεια, οικονομική κρίση, εξωτερικό χρέος είναι προβλήματα τεράστιου βεληνικούς που δεν μπορούν να οδηγήσουν σε περαιτέρω καθυστέρηση της ε, δημοκρατικής ε, ε, διαδικασίας του κράτου δικαίου και το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η επιστροφή στην εξουσία του Πρόεδρου Σελάγια είναι η εκ των ον ουκάνευ προϋπόθεση. Για ένα λεπτό. Η κυρία Λούνατσεκ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σήμερα που μίλησε εδώ πέρα ο Βάτσλαπ Χάβελ για την ελευθερία που κατέκτησε η Ανατολική Ευρώπη πριν από 20 χρόνια, απευθύνομαι σε αυτούς από το ΕΛΚ που λένε να στείλει η Ευρωπαϊκή Ένωση παρατηρητές των εκλογών στην Ονδούρα. Να σας ρωτήσω, τι θα λέγατε εάν πριν από 20 χρόνια η Ευρωπαϊκή Ένωση έλεγε θα στείλει παρατηρητές εκλογών σε μη νόμιμες εκλογέ σε μια δική σα χώρα. Όταν όλοι έλεγαν πως δεν υπάρχει ελευθερία εκεί, πως υπάρχει κλίμα βίας, πως υπάρχει ανασφάλεια. Τι θα είχατε πει τότε, πάνω από 20 χρόνια πριν, εάν λέγαμε ναι, ναι, θα στείλουμε παρατηρητές και όλα είναι εντάξει. Θα λέγατε πως αυτή η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, χάνει την ομοποίησή της με το να στείλει παρατηρητές. Για αυτούς τους λόγους σας ζητώ κυρίες και κύριοι του ΕΛΚ να εφαρμόσετε τα ίδια κριτήρια και στην Ονδούρα. Να μην στείλουμε παρατηρητές σε παράνομες εκλογές. Και ευχαριστώ και την Κομισιόν για το ότι έχει ακριβώς αυτή τη θέση. Ευχαριστώ. Κυρία Επίτροπε, έχετε τον λόγο. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ. Θα είμαι σύντομη. Όχι γιατί δεν αναγνωρίζω τη σημασία του ζητήματος, αλλά γιατί αναγνωρίζω το προχωρημένο της ώρας. Άκουσα με μεγάλο ενδιαφέρον το πάθος με το οποίο τοποθετήθηκαν οι βουλευτές και τις ανησυχίες για την σχέση που πρέπει να έχουμε βράχη πρόθεσμα με την πολύ φτωχή αυτή χώρα που ε, ειλικρινά πρέπει να επανέλθει στην ομαλότητα το συντομότερο δυνατόν. Και την ανησυχία που έχουν συνάδελφοι διαφορετικών αποχρώσεων για τον ρόλο που πρέπει να παίξει η Ευρωπαϊκή Ένωση στις εκλογές και σε εβδομάδες που έρχονται. Σωστή ανησυχία, θα την μεταφέρω και θα συζητήσω με τους συναδέλφους μου. Δεν προξενεί έκπληξη βεβαίω το ότι εγώ θεωρώ εξαιρετικά σημαντικό να συνεχίσουμε να παρακολουθούμε από κοντά την κατάσταση στην Ονδούρα, να ξέρουμε τι συμβαίνει και να λάβουμε τα απαραίτητα μέτρα και να προσφέρουμε στήριξη για να επιληθεί ειρηνικά η κρίση των στομότερων δυνατών. Όπως είπα είναι μια φτωχή χώρα, η επίλυση της κρίσης έχει αργήσει κιόλας και καλωσορίζω την στήριξη των βουλευτών προς την Κομισιόν για τις προσπάθειες που καταβάλουμε για να επιληθεί η κρίση, να παίξουμε και εμείς τον ρόλο μας για να επανέλθει η Ονδούρα στην σταθερότητα των συντομότερων δυνατών. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε. Τελειώσαμε αυτό το σημείο, περνάμε στο επόμενο. Δήλωση της Επιτροπής για το, για το προέλευσης. Το λόγο έχει η Επίτροπος Άστον. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Είμαι ιδιαίτερα ευτυχής που έχω τη δυνατότητα